Προεδρίας του Λουξεμβούργου και καλωσορίζω τον κύριο Ξαβιέ Μπέτλ, Πρωθυπουργό του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Ζων Κέρο. Κύριος Μπέτα, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω έναν απολογισμό απλό όσον αφορά την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Η Προεδρία αυτή, όπως γνωρίζετε, έλαβε χώρα κάτω από δύσκολε συνθήκε, δραματικέ μερικέ φορέ, γιατί η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με πολύ σημαντικέ προκλήσει χωρί προηγούμενο. Κλήθηκε να ανταποκριθεί στην οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Εδώ τα πράγματα πάνε κάπω καλύτερα, βέβαια πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Αστάθεια τόσο στα σύνορα όσο και γενικότερα διότι είναι ένα πρόβλημα το προσφυγικό που παίρνει διαστάσεις τεράστιες στην Ευρώπη. Και άλλα φαινόμενα προσθέθηκαν στο ήδη δύσκολο αυτό πλαίσιο. Είναι ακριβώς η προσφυγική κρίση και η άνοδος της τρομοκρατίας στον κόσμο ολόκληρο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη μετά από τις επιθέσεις που είχαμε στο Παρίσι. Γι' αυτά τα θέματα η Προεδρία αναγκάστηκε να αντιδράσει γρήγορα και συγκεκριμένα. Όσον αφορά την μεταναστευτική κρίση, εδώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τα διάφορα μέτρα ελήφθησαν και στον τομέα ευθύνη των χωρών μελών, αλλά και στο επίπεδο αλληλεγγύης μεταξύ χωρών μελών. Πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε για να υποδεχόμαστε με αξιοπρέπεια τους πρόσφυγες. Πρόκειται για την ε, επανακατάσταση και την μετακατάσταση των προσφύγων. Πρόκειται επίσης για την πολιτική επιστροφή επανεισδοχής, πρόκειται για την καταγραφή τους στα hot spots και πρόκειται και για την ε, ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών μας συνόρων. Όλα αυτά τα μέτρα ελήφθησαν πολύ γρήγορα. Τώρα αρχίζουν να αποφέρουν καρπούς και είναι αναγκαία στα πλαίσια της γενικότερης μεταναστευτική μας πολιτικής, η οποία βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και χαιρόμαστε για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2015. Η εκστρατεία όσον αφορά την μετανάστευση βέβαια θα συνεχιστεί και φέτος. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουμε μέτρα, να εφαρμόσουμε τα μέτρα που έχουμε ήδη αποφασίσει, γιατί με την καλύτερη θέληση των συνομοθετών δεν θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις ροές αν δεν εφαρμοστούν αυτά τα οποία αποφασίσαμε. Είναι κάτι που όλοι το γνωρίζουμε. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του χώρου Σέγγεν, που θα λειτουργήσει μόνον εφόσον τηρούνται οι κανόνες του. Γι' αυτό και από τον Εύρη του 2015 ζητήσαμε να πάμε προς την κοινοτικοποίηση των ε, ελέγχων που γίνονται στα σύνορα. Είναι κάτι αναγκαίο. Δεν μπορεί να αφήνουμε τα κράτη-μέλη να εισάγουν εθνικά μέτρα με τρόπο ασύντακτο. Όλα τα μέτρα που προσφέρει ο χώρος έγκεν δεν χρησιμοποιήθηκαν και πρέπει να γίνει αυτό. Η προτεραιότητα προς το παρόν είναι να κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε σημαντικά τις ροές ε, προσφύγων. Αλλιώς χάνουμε την κοινή μας γνώμη, τους πολίτες μας. Να δούμε τι θα κάνουμε με την ε, μετακατάσταση. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Έγιναν σημαντικές πρόοδες σε αυτό το τομέα, όμως χρειάζονται περισσότερα ακόμα. Και ο καθένας πρέπει να τηρεί τις δικές του υποχρεώσεις και τις δικές του ευθύνες. Είναι θέμα αλληλεγγύης βεβαίως μεταξύ των χωρών μελών. Αλληλεγγύη πολιτική και όχι νομική. Η αλληλεγγύη στην ιστορία της Ευρώπης δεν είναι μονόδρομος. Πρέπει να δίνουμε επίσης και όχι να περιμένουμε μόνο να παίρνουμε. Αλληλεγγύη σημαίνει επίσης συνεργασία με τους εταίρους μας, τα Βαλκάνια και με την Τουρκία. Γι' αυτό και έχουμε το πρόγραμμα δράσης και με τα Βαλκάνια και με την Τουρκία. Παρόλο βέβαια που στην πράξη δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα φιλοδοξίας που έχουμε. Μην ξεχνάμε επίσης το Λίβανο και την Ιορδανία. Οι επιθέσεις που έγιναν στο Παρίσι το 2015 είναι φυσικά μια πολύ κρίσιμη στιγμή και πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία στην Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη, αλλά να μην μπερδεύουμε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία. Πρέπει να φροντίσουμε αυτό το μπέρδεμα να πάψει να γίνεται έτσι εύκολα. Από πλευράς Προεδρίας προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή διάφορα μέτρα ήδη άρχισαν να υιοθετούνται μετά την επίθεση στο Σαρλί Επντό. Δυστυχώ όμως η Ευρώπη δεν αντέδρασε αρκετά γρήγορα. Πρέπει επίσης να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που η οδηγία για το PNR μετά από τρία χρόνια συζητήσεων επιτέλους προχώρησε. Ελήφθησαν επίσης μέτρα γρήγορα και αυτό χάρη στην βοήθεια και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αν προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έγινε χάρη στη στήριξη την επικοδομητική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και δράτω με τι ευκαιρίε αυτή για να σα ευχαριστήσω όλου για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε το τελευταίο εξάμεινο, αλλά και επειδή συνεισφέρατε σημαντικά στην πρόοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορου τομεί που αποτελούσαν και την καρδιά του προγραμματός μας. Αποφασίσαμε σε συναπόφαση διάφορα θέματα και θα αναφέρω κυρίως τον προπολογισμό του 2016. Επίσης ε, υιοθετήσαμε το σύστημα PNR, το ευρωπαϊκό. Επίσης προχωρήσαμε όσον αφορά το τεκμήριο της αθεότητας, την απλοποίηση της κυκλοφορίας δημοσίων εγγράφων, συμφωνία για τους δείκτες αναφοράς και συμφωνεί επίση και για το πακέτο όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Η Λιξεβουριανή Προεδρία οργάνωσε τον πρώτο πολιτικό διάλογο για το σεβασμό και την πρόθεση του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσει που έγιναν του τελευταίου μήνε και εβδομάδε, ακόμα και τελευταίε μέρε, δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η διαδικασία. Είναι ένα διάλογο που μόλι άρχισε. Πρέπει να μπούμε περισσότερο σε βάθος στο διάλογο αυτό. Εσωτερικές υποθέσεις και εδώ χρειάστηκε να έχουμε έκτακτες συνεδριάσεις για να λύσουμε διάφορα ζητήματα, για να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα την κρίση του γαλακτοκομικού τομέα, του χείριου κρέατος και τα προβλήματα της ευρωπαϊκής μεταλλουργίας εξαιτίας της εμπορικής αθέμητης πολιτικής μερικές φορές τρίτων χωρών. Επίσης μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο μηχανισμό διακανονισμού όσον αφορά τους επενδυτές στα πλαίσια της μελλοντικής συμφωνίας TTIP. Και ευχαριστώ τον κύριο Σούλτς, τον πρόεδρο Σούλτς για τη συνάντηση που είχαμε με τους κοινωνικούς εταίρους στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε για το TTIP. Επίσης, τους κοινωνικούς εταίρους από τις 28 χώρες τους βάλαμε γύρω από το τραπέζι για να συζητήσουμε. Για μας το TTIP δεν πρέπει να είναι μια συμφωνία απλώς που θα προσφέρει αξία και εμπιστοσύνη από τους πολίτες θα πρέπει επίσης να αποτελέσει και μια ευκαιρία και έτσι να τη βλέπουμε. Γι' αυτό και πρέπει να προχωρήσει με διαφάνεια και με διαπραγματεύσεις όσο χρειάζεται. Τώρα, στο Ναϊρόμπι η διπουργική συνάντηση ολοκληρώνει το γύρο της Ντόχα. Και εδώ σε πολυμερές επίπεδο είχαμε πρόοδο. Εξυγχρονίσαμε τις μεθόδους εργασίας για την ανταγωνιστικότητα και επικεντρωθήκαμε στην δημιουργία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου υπέρ των επενδύσεων. Και αυτό ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο Juncker. Για περισσότερες ε, επενδύσεις, κάτι το οποίο εγκρίναμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρόκειται για μια γενικότερη αντιμετώπιση του Συμβουλίου που αποτελεί το πρώτο πετραδάκι για την αγορά κεφαλαίων στην Ευρώπη. Επίσης είχαμε την οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους φορολογικούς παραδείσους και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που στέλνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάντα για τα φορολογικά το Συμβούλιο ενέκρινε σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά την πρωτοβουλία BEPS του ΩΣΑ για την διάβρωση της φορολογικής βάσης και την μεταφορά κερδών. Η ευάθεση τώρα στην κοινωνική διάσταση είναι και αυτό κάτι που προχωρήσαμε, μια πραγματική κοινωνική διακυβέρνηση όπως κάνουμε και για τα, τα οικονομικά ζητήματα, έτσι και για τα κοινωνικά. Μετά από πρωτοβουλία του Λουξεμβούργου. Προχωρήσαμε λοιπόν στο τελευταίο εξάμεινο πολύ, αλλά μένουν και πολλά ακόμα να γίνουν. Προχωρήσαμε επίσης όσον αφορά την αηφόρα ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη σε διεθνή φόρα στα πλαίσια της ατζέντα του 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε σε στενή συνεργασία με τους Γάλλους φίλους στα πλαίσια του COP21 στο Παρίσι. Έχουμε μια πρώτη παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Επίσης δουλέψαμε υπέρ της διαφάνειας όσον αφορά την ε, ενεργειακή ένωση στην Ευρώπη και τη βιώσιμη ενέργεια. Ολοκληρώσαμε επίσης το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, εκείνο που έχει να κάνει με την ελευθέρωση των υπηρεσιών ε, μεταφοράς επιβατών μέσω σιδηροδρόμων. Επίσης, ε, ξεκινήσαμε και για τα ψηφιακά, κάτι το οποίο είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέτος ξέρουμε ότι πρόκειται για προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Αγορά. Επιτρέψτε μου εδώ επίσης να εκφράσω και την προσωπική μου ικανοποίηση ως υπουργό ε, Τηλεπικοινωνιών στη χώρα μου για τη συμφωνία που πετύχαμε με τους συνομοθέτες για την πρόταση οδηγίας που θα ενισχύσει την ασφάλεια των ψηφιακών ε, δικτύων και δικτύων πληροφοριακής στην Ευρώπη. Βέβαια πολλά μένει να γίνουν ακόμα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε και την ε, Ασία. Πολλοί νέοι, νέα ταλέντα, με σημαντικά προσόντα ανακάζονται να φεύγουν από την Ευρώπη και να πηγαίνουν αλλού επειδή στην Ευρώπη έχουμε 28 διαφορετικές ρυθμίσεις. Η συνεργασία λοιπόν, Πρόεδρε, ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σα πω ότι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την Προεδρία μα. Πετύχαμε για τον προπολογισμό πέντε μέρε πριν τη λήξη τη προθεσμία να συμφωνήσουν τα δύο όργανα και οι τρεις μαζί φροντίσαμε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να λειτουργούμε πιο αρμονικά και να νομοθετούμε καλύτερα. Και πετύχαμε πολιτική συμφωνία από το Δεκέμβριο και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα εφαρμοστεί αφού αποφανθεί την άνοιξη το δικό σας σώμα. Θέλουμε να εξυγχρονίσουμε επίσης την νομοθετική διαδικασία για τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια αλλά και λιγότερο διοικητικό άχθο όσον αφορά τον προπολογισμό, γιατί είναι πολύ βασικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, μικρέ και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτού του καιρού κρίσης που ζούμε, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε με το ευρωπαϊκό όνειρο και να σκεφτούμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε μπροστά μας τις νέες γενιές. Πρέπει να μην ξεχνάμε το σχέδιο ερήνευσης με το οποίο ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την τύχη να είμαι από το Λουξεμβούργο. Έχω σπουδάσει στη Γαλλία, έκανα εράσμου στην Ελλάδα. Και πρέπει να σα πω ότι ανακάλυψα κάτι το οποίο αν είχα γεννηθεί αργότερα δεν θα είχα διαπιστώσει. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη φοιτητή και πήγα στα Σκόπια με το αυτοκίνητο και είδα ότι υπήρχαν κλειστά σύνορα. Με ελέγχου έπρεπε να σταματήσω ξανά και ξανά στα τελωνία, να βρω κλειστά τελωνία, πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουν οι σημερινές γενιές, να σταματήσω για συνάλλαγμα κλπ. κλπ. Όλα αυτά όμως δεν υπάρχουν πια. Τώρα έχουμε ένα χώρο ελευθερίας. Μπορούμε να ερωτευτούμε κάποιον χωρίς να χρειάζεται διαβατήριο. Είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίζουμε αυτό καθημερινά και κυρίως τις νέες γενιές να ξέρουν γιατί αγωνιζόμαστε. Από πλευρά τη χώρα μου, λοιπόν, είναι πήγον να συνεχίσουμε προ την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γιατί εκεί βρίσκονται οι λύσει τη κρίση που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ, σίγουρα πολλά περισσότερα θα μπορούσα να σα πω, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Η χώρα μου είναι ευτυχή που μπόρεσε για δεύτερη φορά να αναλάβει την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίστηκε στην ε, δικιά σα στήριξη. Σα ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστώ και όλου του υπαλλήλου, είτε από τη δικιά σα την πλευρά, είτε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την πλευρά του Λουξεμβούργου για το έργο του. Εκείνοι δούλεψαν σκληρά για να μπορέσουμε με τόσο καλό τρόπο να πετύχουμε τους τελευταίους έξι μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ και το λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος Επιτροπής κύριος Γιονκέρ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρωθυπουργέ, από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε διαπράχθησαν νέες φρικαλαιότητες στην Κωνσταντινούπολη και την Τσακάρτα. Η δημοκρατία μας που εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο και οι αξίες που αποτελούν τα θεμελιά της είναι πολύ πιο ισχυρές από αυτές τις τρομοκρατικές πράξεις. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και η τρομοκρατία που ελοχεύει δεν πρόκειται ποτέ να μας εκφοβήσει θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διαφυλάξουμε τις ελευθερίες μας, τον τρόπο ζωής μας, την, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε όλοι μαζί και εν ολίγης ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ως προς την Λουξεμβουριανή Προεδρία, κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά θα πρέπει να πω ότι πρέπει να αποτίσουμε φορό ε, στο Λουξεμβούργο σε όλο το επιταλείο της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς που τον συνόδευσαν. Η Προεδρία έκανε πολύ καλή δουλειά. Και στην περίπτωση του Λουξεμβούργου αυτό πάντοτε επαληθεύεται. Η ουσία είναι πάντοτε όχι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα. Αξιοσημείωτη ποιότητα αυτής της Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Κάτι που συνέβη και παλιότερα. Το 1985, θυμηθείτε, η Προεδρία του Λουξεμβούργου προέβλεψε την ενιαία πράξη που σημάδεψε τη γέννηση της εσωτερικής αγοράς και η διακυβερνητική συνέλευση για την οικονομική Ένωση έγινε επί Λουξεμβουργιανής Προεδρίας στη δίκαιο το 1997. Οι πρώτες συζητήσει για, για τη διεύρυνση που επέτρεψαν στην Ευρώπη να ανασένει με τον ίδιο ρυθμό το ίδιο και για την τωρινή κυβέρνηση που ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Αποδείχτηκε αντάξια των προσδοκιών μας. Η Προεδρία αυτή ασκήθηκε σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσκερής. Πρώτα απ' όλα με το ζήτημα της μετανάστευσης. Με ένα διάλογο επικοδομητικό μεταξύ 28 διαφορετικών εθνικών πραγματικότητων και με απόψεις κάποιες φορές αντιδιαματρικά αντίθετες. Για κάποια βασικά ζητήματα για τα μητρώα των επιβατών των αερομεταφορών και για άλλα ζητήματα που βρίσκονταν στο νεκρό σημείο μέχρι τώρα επετεύχθη και η διακυβερνητική συμφωνία που αναφέρατε είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητούμε ούτε τη σημασία ούτε το εύρος. Η κομψότητα με την οποία η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου καθοδήγησε τις συζητήσει, τις συζητήσεις, τις τεχνείς συζητήσεις για το κλίμα στο Παρίσι ήταν μια επίδοση που δεν αναφέρεται συχνά αλλά παραμένουν στο πρόσφατο ιστορικό επιτυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την κρίση των προσφύγων. Ε, με την φωτισμένη καθοδήγηση του Υπουργού ε, του Λουξεμβουργού και τη βοήθεια και του Κοινοβουλίου βρήκαμε συμφωνία ε, σε επίπεδο πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση και το μετατοπισμό των μεταναστών. Και πολλά από αυτά έλαβαν και σάρκα και οστά, δεν παρέμειναν μόνο κενό γράμμα. Επίσης, επιτελέσαμε πρόεδρο και για άλλα θέματα. Ίσως αργά για το γούστο κάποιον, όπως τη λειτουργία των πρώτων hot spot, ή την ε, εξασφάλιση της οδού των Βαλκανίων, ένα πρόγραμμα συνεργασίας με την Τουρκία και με τη βοήθεια της Προεδρίας είχαμε και την απαραίτητη χρήσιμη συνεργασία με τους Αφρικανούς μας εταίρους. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη διάθεσή μας νέα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε, για να πετύχουμε μάλλον μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και δραστικότητα την κρίση ε, των προσφύγων. Θα πρέπει να προβλέψουμε και άλλα εργαλεία, όπως την προστασία των κοινών εξωτερικών μας συνόρων ή τη δημιουργία ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής. Η μετανάστευση είναι, ε, και η αντιμετώπιση του όλου ζητήματος είναι ένα μακρόπνο εγχείρημα. Θα πρέπει να μην εφησυχάσουμε, αλλά να συνεχίσουμε το έργο που η Λουξεμβουργιανή Προεδρία ε, ξεκίνησε με τόσο εύστοχο τρόπο. Hotspot, κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Σύνοριο Φυλακή, όλα αυτά τα στοιχεία συμβαδίζουν. Δεν μπορούν να ε, αντιμετωπιστούν το ένα ξεχωριστά από το άλλο. Όλα αυτά τα μέτρα από κοινού θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές και τους κινδύνους που μπορεί να απειλούν το χώρο του Σέγγεν. Οι απειλές αυτές είναι σημαντικές. Μπορεί να είναι και η ίδια επιβίωση του Σέγγεν που διακυβεύεται. Σήμερα, ατάκτος, προβλέπονται και πάλι έλεγχοι στα σύνορα, αλλά θα αντιληφθούμε ότι το οικονομικό κόστος είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή. Αύριο κιόλα. Και μεθαύριο θα αναρωτηθούμε γιατί είχαμε οικονομική ένωση όταν δεν έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά. Και κατά συνέπεια θα γνωρίσει απειλές κατά των ίδιων των θεμελίων της Ευρωπαϊκή Ένωση. Χειρότερες από αυτές που σήμερα μας βαραίνουν. Με όλα αυτά τα προβλήματα η Λουξεμβουργιανή Προεδρία διαχειρίστηκε τα της Προεδρίας της με μεγάλο θάρρος γιατί δεν έχανε ποτέ και την ευρύτερη εικόνα. Υπήρχαν πολλά ζητήματα, πολλά ζητήματα προς διαπραγμάτευση. Ζητήματα όπως ε, αυτό των δεδομένων επιβατών πτήσεων. Η βασική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που είναι μια ιστορία λουξεμβουριανή γιατί το 2012 η κυρία Ρέντινγκ έκανε τις σχετικές προτάσεις για τον κανονισμό μια λουξεμβουριανή προεδρία ξεκίνησε την ιστορία και μια Λουξεμβουρ... ένας λουξεμβουριανός μάλλον πρόεδρος επιτροπής έκανε δεκτές τις προτάσεις και μια λουξεμβουριανή προεδρία κατέληξε στην πρόταση που εγκρίθηκε. Μια λουξεμβουριανή υπόθεση λοιπόν και χαίρομαι ιδιαίτερω και θέλω να ευχαριστώ και τον Πρωθυπουργό για την ε, συνεργασία. Αυτή η Προεδρία πιστεύω ήταν μια επιτυχημένη Προεδρία. Δεν υπάρχει καμία κανένας ψόγος που θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε στην, προς την Προεδρία του Λουξεμβούργου επέτυχε πολλά πράγματα. Κάνατε πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Ρέντινγκ. Κύριε... Πρόεδρε, οι μικρέ χώρε είναι σε θέση να φέρουν ει πέρα πολύ καλά τα εξάμενα τη Προεδρία. Το απέδειξε το Λουξεμβούργο και άλλη μια φορά, διότι είχε την θεσμική εμπειρία ε, από δεκαετίε κιόλα. Βεβαίω, ο χαρακτήρα τη Προεδρία έχει αλλάξει από τη συνθήκη τη Λισαβόνα που υποκατέστησε τι χιλιόμενε Προεδρίε από την μόνιμη Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βεβαίω, χρειάστηκε να υπάρξει και διαπραγμάτευση ανάρθρο και χάρη σε αυτό το πλέον ε, το έργο των λουξεμβουριανών ε, συνεργατών επέτρεψε να επιτευχθεί πρόοδος σε δεκάδες θέματα. Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η διαθεσμική συμφωνία, το πακέτο μετρών για, για τους σιδηροδρόμους, το Μητρό Επιβατών και ούτω καθεξής. Ήταν ένα έργο το οποίο ε, μπορούσε να χειριστούν κατάλληλα λουξεμβουργιανοί με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα. Οι συνεργάτες του Λουξεμβούργου και όσοι του στήριξαν ήταν ε, πολυάριθμοι και πραγματικά τους ευχαριστούμε. Η κυβέρνηση μπόρεσε να προωθήσει πολλά θέματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ε, βρέθηκε σε μια από τις πρώτες θέσεις η ε, δράση του σημειώθηκε, όπως και η δράση του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων του κ. Σμιτ, ήδη στην COP21 ε, όπου η Προεδρία του Λουξεμβούργου επένεσε την ε, Γαλλία για το εξαιρετικό της έργο και κάνοντας την Ευρώπη να μιλήσει με μια ενιαία φωνή. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε όλες και όλους. Κατά τα άλλα αντιμετωπίσαμε κρίσεις άνευ προηγουμένου και άνευ χωρίς τέλος. Ήδη αυτό το σκοτεινό, αυτή η σκιά που έπεσε στην Ευρώπη από τις μεταναστευτικές ροές και τους πρόσφυγες, η άνοδος των εθνικισμών και των εγωισμών, η απειλή κατά του κοινού μέλλοντος της Υπήρου μας, αυτά τα σοβαρά προβλήματα ε, δεν είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπίσει μία μόνο προεδρία. Πρέπει να τα ξεπεράσει και οι κρίσεις παραμένουν. Το 2016 θα πρέπει να είναι ένα σημείο καμπή στις ιδρυτικές γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται συνοχή, σεβασμός, αλληλεγγύη και μια Ευρώπη που να προχωρά, να προοδεύει. Αυτό θέλουμε να συμβεί. Ευχαριστώ εκ μέρους της Δημοκρατικής Ομάδας, ε, η κυρία Τελβού. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι ως ε, Λουξεμβούργια, σοσιαλίστρια, δεν θα φανταστεί κανείς ότι θα πω κάτι κακό για την Λουξεμβουριανή Προεδρία, θα την επενέσω ασφαλώς. Και ως Ευρωπαία θέλω να επενέσω την Λουξεμβουριανή Προεδρία για το τελευταίο εξάμεινο. Ενώ η Ευρώπη αντιμετώπιζε, όπως αντιμετωπίζει ακόμη τεράστιες προκλήσεις, χρειάστηκε να διαφυλαχθούν οι κοινέ μας αξίες, αυτές που αποτελούν και την ουσία ύπαρξης της Ένωσης. Ο κύριος Άσομπορν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες, ταξίδεψε παντού. Ο Νικόλα Σμιτ διανυκτέρευε εδώ στην Ολομέλεια, στο Κοινοβούλιο. Τα κάνατε πολύ καλά. Πάνω από όλα όμως, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δουλειά που έγινε στις λιγότερο θεαματικές, στα λιγότερο θεαματικά θέματα. Δεν θα τα εκθέσω όλα, αλλά είναι δουλειά σοβαρή και διακριτική που έγινε για χρόνια. Η συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ήταν επίσης υποδειγματική. Αυτό ασφαλώς οφείλεται στην προσήλωση της Λουξεμβουργιανής κυβέρνησης, αλλά πολύ περισσότερο και στην προσήλωση των υπαλλήλων του Λουξεμβούργου και εκείνων που βρίσκονται εδώ στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη αντιπροσωπεία και θέλω ιδιαίτερως να εκφράσω προς αυτούς προς τις ευχαριστίες μου. Το μόνο που μένει είναι να εκφράσω την ευχή οι επόμενες προεδρίες να δείξουν την ίδια καλή διάθεση συνεργασίας, την ίδια προσήλωση και την, το ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης για την Ένωση που το έχει τόσο ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντελβού, ομάδα συντηρητικών μεταρρυθμιστών, κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα θέματα της ασφάλειας ήταν ψηλά στην ατζέντα της Λουξεβουργιανής Προεδρίας και σωστά επετέχθη μία συμφωνία στον τομέα του PNR, των στοιχείων των επιβατών, κάτι που περιμέναμε πολλά χρόνια και έτσι τώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Κατά της τρομοκρατίας επίσης αγωνίστηκε η Ευρώπη σε διάφορα επίπεδα. Στο να μπορεί να βρει τους τζιχαντιστές στο διαδίκτυο, για παράδειγμα. Πετύχαμε επίσης συμβιβασμούς σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με στην αστυνομική συνεργασία. Στο θέμα των προσφύγων δεν έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα. Οι πρόσφυγες προσπαθούν να φτάσουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ανατολικές χώρες στην Ευρώπη πρέπει να αναλάβουν και αυτές όμως τις ευθύνες τους. Για να διαφυλάξουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται μια συστηματική πολιτική. Πρέπει να σταματήσουν επίσης οι ροές νέων προσφύγων και αυτό θα γίνει αν συστηματικά αποθούμε τους λαθροδιακινητές. Για εκείνους που ζητούν άσυλο και περνάνε μέσα από χώρες transit δεν πρέπει στην Ευρώπη να ζητούν άσυλο. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να λύσει όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε τι αριθμό ετούν τον άσυλο θα δεχτούμε και πόσους μπορούμε να υποδεχτούμε. Έτσι, έχοντας αποφασίσει κάτι τέτοιο και θέτοντας το σε εφαρμογή, αποθούμε τους λαθροδιακινητές. Θέλω επίσης να πω ότι δεν μας είπατε, δεν αναφερθήκατε καθόλου στο θέμα του Brexit. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα, εκ μέρους των φιλοθερών ο κύριος Γκέρενς. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, όταν παρουσιάσατε τι προτεραιότητε τη Προεδρία σα, πολλοί από εμά σα είπαμε ότι έξι μήνε τη Λουξεμβουργενής προεδρία θα ταυτιζόντουσαν με μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και επισφαλή για την Ευρώπη. Υπήρχαν ήδη κρίσεις στην Ευρώπη τον Ιούλιο και έγιναν υπαρξιακές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια. Έγιναν υπαρξιακές γιατί οι χώρες μας δεν είναι έτοιμες να τιμήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέσα που χρειάζεται για να λύσει τις κρίσεις αυτές. Επίση, πρέπει να πω ότι η Προεδρία σα κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλέ σημαντικέ προκλήσει. Προπολογισμό του 2016, για παράδειγμα, που βέβαια τζιματζίμα καταφέραμε να τον εγκρίνουμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Είχαμε επιτυχίε και σε θέματα εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνη. Η Προεδρία Επίσης, συνεισέφερε για να προχωρήσει το θέμα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ακόμα πρόθυσε και θέματα στον τομέα της γεωργίας. Όμως έπρεπε να αποδείξουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και αν δεν ήταν σίγουρα από πριν ότι θα πετύχουμε και κάνατε προσπάθειες. Όμως, ορισμένες χώρες μέλη επιβραδύνουν τα αποτελέσματα και δεν δείχνουν αλληλεγγύη όπως το θέμα των προσφύγων. Πολλές χώρες μέλη αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αφήνουν σε άλλους να αναλάβουν τις ευθύνες όλων. Τρεπόμαστε συχνά που βλέπουμε ότι οι ορισμένες χώρες αμφισβητούν αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως εκείνες του Σέγγεν. Μήπως χρειάζεται ομοιοπαθητική για να λυθεί το πρόβλημα αυτό των ετούντων άσυλο. Η Γερμανία σήμερα 24.000 υποδέχεται και άλλες χώρες αντίστοιχα νούμερα σε μία περίοδο δύο ετών. Στις αρχές του 2016 είμαστε σε κρίση αλληλεγγύης. Το ότι δεν μπορούμε να μοιραστούμε τις ευθύνες μας μεταξύ των 28 δεν είναι βέβαια καθόλου θετικό. Το Λουξεμβούργο είναι βέβαια χώρα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση. Βασιζόμαστε σε εσά ε, στο ταλέντο σας, στη, στο προσωπικό σας, στην εμπειρία που έχετε για να προχωρήσει περισσότερο η Ευρώπη και το ίδιο και για την επόμενη Προεδρία. Πρέπει να ξεπεράσουμε το διακυβερνητικό, διότι παραλύει την Ευρώπη και επιτρέπει στους εθνικιστές να εξέχουν. Η Ευρώπη αξίζει κάτι καλύτερο και οι πολίτες της αξίζουν μια Ευρώπη με αλληλεγγύη και αποτελεσματική. Δεν πρέπει να παραμείνει όνειρο. Για αυτούς που παραμένει όνειρο πρέπει να πω ότι δεν θα είναι όνειρο αλλά πραγματικότητα εάν όλοι αποφασίσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία ο κ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπέτελ, κύριε Γιουνκέρ, λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να συμμεριστώ ούτε εγώ ούτε η πολιτική μου ομάδα την αισιοδοξία, του επένους, την αυρότητα ανάμεσα σε Λουξεμβουριανούς. Η Λουξεμβουριανή Προεδρία προσπάθησε, αλλά τώρα μετράμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου μετά από ένα εξάμεινο έργο και οι αριθμοί και τα γεγονότα επιβάλλουν ανησυχία εγρήγορση ευθύνη και όχι αυταρέσκεια. το σεπτέμβριο αποφασίσατε τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων με αναλογική κατανομή σε όλη την ευρώπη. ποιος είναι ο απολογισμός; μερικές εκατοντάδες άνθρωποι ούτε καν 1% υλοποίηση των αποφάσεων. αφήσατε την ελλάδα μόνη και ουσιαστικά αβοήθητη να σηκώνει το, 85% των προσφυγικών ροών. Υπογράψατε μια συμφωνία πλαίσιο με την Τουρκία, αλλά ο κύριος Τίμερμανς λέει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην μείωση των προσφυγικών ροών, γιατί οι τουρκικές αρχές περιμένουν τα λεπτά χωρίς να υλοποιούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Και μέσα σε αυτό το έδαφος των εγωισμών των εθνικισμών της ξενοφοβίας φουντώνουν κραυγές μας φταίει σέγγεν μικρότερη σέγγεν σημαίνει καθόλου σέγγεν και κατάρρευση της σέγγεν σημαίνει κατάρρευση της ευρωζώνης και αυτό δεν θα κοστίσει μόνο στη δημοκρατία ή στους πρόσφυγες θα κοστίσει πανάκριβα και στην οικονομία. επειδή λοιπόν αυξάνεται και η ανεργία και η φτώχεια και η οικονομική ανάπτυξη είναι ασθενική είναι η ώρα όχι να συγχαίρεστε μεταξύ σας αλλά να πάρθουν μεγάλες πρωτοβουλίες ταυτόχρονα για την αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων ανάπτυξη με καταπολέμηση της ανεργίας και αντιμετώπιση του προσφυγικού με ενιαίο ευρωπαϊκό τρόπο. ευχαριστώ. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Αξιότιμη ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρωθυπουργέ Μπέτλ οι πρωθυπουργοί σας, όπως όλες, απαρτίζεται από σχέδια και επιτεύγματα. Ούτε για τα σχέδια είσαστε μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος, ούτε για τα επιτεύγματα. σε σχέση με τα όσα είχαν σχεδιαστεί και τα όσα υλοποιήθηκαν, ε, βλέπω κάποια σημεία στα οποία δεν βλέπω να έχετε πολύ σοβαρή επιτυχία, όπως ένα νέο απολογισμό ισορροπίας μεταξύ ε, ε, εμπορικής και οικονομικής πολιτικής, την οικολογική στροφή στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η θετική όμως επίδοση νομίζω το, γενικό πρόσημο είναι θετικό και βέβαια σε σχέση με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων βλέπω να έχετε καταλήξει ένα καλό αποτέλεσμα. Η δική σας ε, η προσφορά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, η δική σας η προσωπική αλλά και ε, όλου του, ε, του Υπουργικού Συμβουλίου κυρίως σε σχέση με την διάσκεψη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή ήταν πολύ επιτυχημένη και σας ευχαριστώ ρητά γι' αυτό. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι στην Ευρώπη επαναρχόμαστε σε μια ομαλότητα εκ νέου. Η ομαλότητα αυτή είναι μια σόρευση κρίσεων και απειλών και δεν φαίνεται να αλλάζει σύντομα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες, άντρες και γυναίκες, αυτούς που φοβούνται ότι θα χάσουν την ασφαλεία τους, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχία. Η πρόκληση δεν έχει μόνο ρητορικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για hope and change. Πρέπει και να υλοποιούμε αυτό που χρειάζεται ο πολίτης για να φέρουμε την πραγματική αλλαγή. Θα δούμε αν θα υλοποιηθούν αυτές οι αλλαγές λοιπόν. Είχατε πει στην αρχή της Προεδρίας σας ότι πρέπει να εισακούονται οι πολίτες, πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον πολίτη. Για μένα ήταν κεντρική σημασία σε αυτή η φράση. Για μένα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακούω τον πολίτη και να τον αφουγκράζομαι, ακόμα και εκεί που δεν λέει αυτό που θέλει να πει. Όταν λέτε κύριε Μπέτλ ότι πρέπει να αλλάξει όταν λέγεται με αλφαγιώτο ότι πρέπει να αλλάξει τη TIP, σημαίνει να αφογκραστούμε τον πολίτη που έχει πολλές επικρίσεις και ενσυχίες σχέση με το TTIP. Άλλωστε μας το λέει και η Eurostat και να αλλάξουμε. Στην αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη δεν σημαίνει να απαιτούμε εμείς μόνο, αλλά να ακούμε και αυτό που περιμένουν ως αλληλεγγύη οι άλλοι. Το να μιλούμε για να μιλούν οι Πολωνοί για αλληλεγγύη σε σχέση με το προσφυγικό σημαίνει ταυτόχρονα πρέπει να τους δώσουμε και μία αλληλεγγύη ως προς το North Stream. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε τη διαφύλαξη της Ευρώπης των εθνών και τα ευρωπαϊκά έθνη. Τον κίνδυνο να ξαναγυρίσουμε σε μια κατακαιρματισμένη Ευρώπη, στον κίνδυνο ενός Brexit. Πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική ευρωπαϊκή, μια στρατηγική εθνική, γιατί μέχρι στιγμής ευρωπαϊκή λύση είναι μόνο αυτή την οποία υποστηρίζει η Γερμανία. Εάν λοιπόν επιβάλλεται πάντα η βούληση της Γερμανίας, αυτό θα είναι και η καταστροφή της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Βαλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σήμερα ζούμε ένα πολλαπλό παράδοξο της Ευρώπης με του Λεξομποριανή Προεδρία που ακριβώς ε, μιλά για μεγάλες επιτυχίες σε επίπεδα δικαιοσύνης και φορολογικής διαφάνειας. Μιλάμε, μιλάω για την περίπτωση της αντάλλαγη, ε, ανταλλαγής πληροφοριών, την περίπτωση των φορολογικών ε, συμφωνιών, των tax rulings. Γιατί δεν λέγεται ότι είναι τελείως περιορισμένο το μέτρο αυτό και τελείως μη φιλόδοξο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Γιατί δεν μιλάμε για την υπόθεση για την οποία η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεωρήσει ότι υπάρχει παράνομη κρατική ε, ρύθμιση από την πλευρά του κράτου του Λουξεμβούργου. Και ω προ του φορολογικού παραδείσου, ε, το Λουξεμβούργο θα είναι μία από τι χώρε ε, που σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν τον τομέα κάνουν ακριβώ αυτό που του συμφέρει, σε αντίθεση με την Ιταλία και τι υπόλοιπε χώρε. Οι αποφάσει των Βρυξελών επικρίνονται πολύ συχνά και δημιουργούν αβεβαιότητα για τι επιχειρήσει, δείχνοντα τον πραγματικό πρόσωπο του Λουξεμβούργου. Μπορείτε λοιπόν να συνεχίσετε να λέτε παραμύθια μεταξύ σα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα μια χώρα που επί χρόνια έχει ευημερήσει στι πλάτε των Ευρωπαίων εταίρων, ε, κλέβοντα ε, νόμιμε θέσει εργασία από άλλου που πλήρωσαν οι πολυεθνικέ. Και όπως είπε η Προεδρία και ο Πρόεδρος Γιούνκερ, ε, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες στην Επιτροπή Τάξε για να μας ε, πείτε τι άποψη έχετε για την έκθεση Κριτικέ και την πρόσκληση αυτή τη στηρίζουν και δύο μεγάλε ομάδε. Ελάτε λοιπόν να αντικρούσετε αυτέ τι κατηγορίε, ιδάλω δεν θα είστε άξιοι να έχετε λάβει όλου αυτού του επένου. Ευχαριστώ κύριε Λεπέν. Κύριε Πρωθυπουργέ του Λουξεμβούργου, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, η Λουξεμβουργιανή Προεδρία ξεκίνησε με αποκαλύψει για το LuxLeaks. Η μέθοδοι δηλαδή υπέρ των πολυεθνικών που ήταν οργανωμένες οι μέθοδοι αυτές από το Λουξεμβούργο. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν κάποια στιγμή να το θάψουν το θέμα και αρνήθηκαν να υπάρξει ερευνητική επιτροπή. Ησυχία. Εδώ με ξαπατούμε. Και για τα θέματα τα φορολογικά όλα καλά. Μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν περισσότερα και φορολογούμενοι, γιατί το Λουξεμβούργο και άλλοι φορολογικοί παράδοση οργανώνουν τέτοιες μεθόδους φοροποφυγής. Και λίγη η Προεδρία του Λουξεμβούργου με τη δραματική κατάσταση των προσφύγων, που παίρνει τεράστιες διαστάσεις εξαιτίας του αριθμού των ανθρώπων που έρχονται προς την Ευρώπη και τεράστια εξαιτία και των ε, επιθέσεων των σεξουαλικών που έγιναν ε, στην κολονία. Αυτές οι σεξουαλικές επιθέσεις δείχνουν ότι ο πολιτισμός μας οπισθοχωρεί, πάει πίσω. Όλοι πρέπει να υποστηρίξουμε την ελευθερία των γυναικών να κυκλοφορούν ελεύθερα στις πόλεις. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες, οι οποίοι συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτό πρέπει να πάψει. Η χώρα μου φέτος υπέστη πολλά δράματα. Οι τρομοκρατικές ισλαμιστικές επιθέσεις επανελήφθηκαν ξανά και ξανά. Η καταπολέμηση του Ισλαμισμού και ο έλεγχος των συνόρων μας είναι κάτι αναγκαίο για να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας. Χρειάζεται όμως ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή. Τα έθνη διαλύονται. Πρέπει να τα στηρίξουμε, να τα διαμορφώσουμε. Ο Η πολυπολιτισμική διάσταση ε, χωρίζει τους ανθρώπους, τους διαλύει. Πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να επιστρέψουμε σε το δικό μας πολιτισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσο, μία εγγεγραμμένος βουλευτής. Κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορεί κανείς να αναμένει η εκάστοτε Προεδρία να επιλύει κάθε πρόβλημα. Μπορεί όμως και οφείλει να αναμένει να δώσει σωστές κατευθύνσεις για όλα τα προβλήματα. Ένωση για τους πολίτες ήταν το σύνθημα. Δηλαδή ο πολίτης έπρεπε να ενταχθεί, να μπει στο επίκεντρο της προσοχής των πολιτικών μας. Αυτό δεν επιτεύχθη δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες και οι ανάγκες των πολιτών. Η δε μεταναστευτική κρίση δείχνει ότι αυτή η πολιτική ελίτ απέχει πολύ από τις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών. Αποφασίστηκε να ρυθμιστεί το σύστημα με ένα με μια κανονιστική παρέμβαση, με ποσοστώσεις. Δεν δόθηκαν απαντήσεις όμως ε, στους προβληματισμούς των πολιτών. Και εδώ είναι μεγάλη και βαριά η ευθύνη. Εκατοντάδες χιλιάδες ε, πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη και απειλούν την ε, κουλτούρα της. Επίσης αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Τουρκία η οποία υποτίθεται ότι θα διέκοπτε τις μεταναστευτικές ροές. Ούτε αυτό επιτεύχθη. Σε σχέση με τη Ρωσία και χρονικά και ε, ως προς το φάσμα τους επεκτάθηκαν και παρατάθηκαν οι κυρώσεις, χωρίς αυτό όμως να αποδυναμώσει τον Πούτιν. Ταυτόχρονα πολλές ήταν οι επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη που υπέστησαν βαρύτατα πλήγματα. Όλα αυτά συνιστούν αποτυχία. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Κέιλαμ. Το Λουξεμβούργο ανέλαβε την Προεδρία τη στιγμή της μεγαλύτερης κρίσης για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όμως δεν κλονίστηκε. Ε, παρέμεινε σταθερό και με επαγγελματισμό, αξιοπιστία και κομψότητα ανέλαβε τα ηνία. Και εσείς κύριε Γιούνκερ ακολουθήσατε αυτή την μακρόχρονη παράδοση επάξια. Ένα σύγχρονο κράτος είναι καλό να μπορεί να μιλήσει με μια ε, φωνή σταθερότητας. Η Εστονία είναι ε, πολύ πρόθυμη να διδαχτεί από την εμπειρία του Λουξεμβούργου που έχει μεγάλη θεσμική εμπειρία. Τρει παρατηρήσεις. Πρώτον, ω προ την ε, κυβερνοασφάλεια υπήρχαν ε, μεγάλες, μεγάλα επιτέγματα. Πρώτα απ' όλα η συμφωνία για την ε, σχετική οδηγία και το πακέτο μέτρων για την προστασία δεδομένων. Και τα δύο είναι η ραχοκοκαλιά όχι μόνο τη κυβερνοασφάλεια αλλά και τη ε, ολοκλήρωση τη ψηφιακή ένωση στην Ευρώπη. Έπειτα, ε, εκφράζω την ικανοποίησή μου που επί Λουξεμβουργιανή Προεδρία προβλέφθηκαν κυρώσει για να αντιμετωπιστεί η επιθετική στάση τη Ρωσία και σε σχέση με όσα συμβαίνουν με το Ισλαμικό κράτο στην Συρία. Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρηθούν οι κυρώσει αυτέ μέχρι οι συμφωνίε του Μίνσκ να ε, υλοποιηθούν πλήρω. Και έπειτα είναι πολύ θετικό που το Συμβούλιο στήριξε την απλούστευση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που προβλέπει ευκολότερη πρόσβαση ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης έγιναν απόπειρε για απλοποίηση των κανόνων της κοινής αγροτικής πολιτικής, όμως η μέγιστη πρόκληση είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κοινέ αγροτικέ πολιτικέ με την πραγματική έννοια του όρου, αλλά υπάρχουν 28 εθνικέ γεωργικέ πολιτικέ με κοινό παρονομαστή ότι όλοι θέλουν πόρου και κονδύλια από τον ίδιο κορβανά. Γι' αυτό συνεχίζονται τα σφάλματα και οι ελλείψεις. Και αυτό θα απασχολήσει και την επόμενη Προεδρία. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στο Λουξεμβούργο. Κύριο Ζάντ, Σοσιαλιστική Ομάδα. Στο δεύτερο ημίση του 2015 η Λουξεμβουργιανή Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξαν μεγάλη αποφασιστικότητα και προσπάθησαν να καθοδηγήσουν την Ευρώπη εκτός ε, των ε, ταραγμένων νερών της κρίσης. Ωστόσο η ελληνική κρίση, η προσφυγική κρίση ήταν ε, όλες κρίσεις που αντιμετωπίστηκαν με πυροσβεστικό τρόπο. Δυστυχώς έδειξαν τα γεγονότα ότι δεν ισχύουν οι υποθέσεις και προϋποθέσεις που θεωρήθηκαν δεδομένες. Έχουν αλλάξει οι πραγματικότητες σε σχέση με το παρελθόν. Τα αποτελέσματα των εκλογών του τελευταίου εξαμήνου δείχνουν οι πολίτες το έχουν αντιληφθεί αυτό. Είναι προφανές ότι όταν κάνει κανείς πυροσβεστικές παρεμβάσεις δεν μπορεί να μειώσει τα προβλήματα. Βεβαίως υπάρχουν ενδείξεις ε, ότι χρειάζονται νέε στρατηγικές, ότι χρειάζεται να μελετήσουμε, να αναθεωρήσουμε τις υποθέσεις μας και τις ε, μεθόδους, όχι τα ε, οράματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Και πρέπει να κοιτάξουμε μια νέα πολιτική συνοχή στην Ευρώπη, την πολιτική για τη μετανάστευση, τι συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση, το μείγμα κρατικού και δημόσιου τομέα και βέβαια τη δημιουργία θέσεων εργασία. Κύριε κύριος Κέρκοπ. Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γιούγκερ, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας όσον αφορά τη συμφωνία για τα στοιχεία επιβατών. Είναι σε καιρούς τέτοιων προκλήσεων κάτι πολύ σημαντικό που το πετύχαμε. Δεν χρειάζεται περισσότερη καθυστέρηση για να εγκρίνουμε τα εφαρμοστικά μέτρα η ελευθερία μας, η ασφάλειά μας διακυδεύεται εδώ. Μιλάω και ως εισηγητής για τον ε, μηχανισμό μετεγκατάστασης. Το Δουβλίνο έχει ξεπεραστεί. Φυσικά και χρειαζόμαστε νέες ιδέες σε ένα τόσο πολύπλοκο θέμα και χρειάζονται και συμβασμοί. Γι' αυτό και πιέζονται την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε, να εφαρμόσουμε καταρχήν αυτά τα οποία διαθέτουμε πολλά από τα προβλήματά μας έχουν να κάνουν με το ότι δεν τηρούνται σημερινοί κανόνες και γι' αυτό υπάρχουν συνέπειες. Νόμοι χωρίς εφαρμογή δεν έχουν νόημα. Ελπίζω λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτό τους επόμενους μήνες, στην εφαρμογή δηλαδή των όσων ήδη έχουμε. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Γκουετόρ, κύριος Χουντής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, κύριε Πρωθυπουργέ του Λουξεμβούργου, αντικειμενικά και η δική σας Προεδρία έχει ταυτιστεί όχι μόνο για τους έλληνες αλλά και όσους πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή ένωση είναι ένας χώρος δημοκρατίας έχει ταυτιστεί λέγω με την επιβολή πολιτικού πραξικοπήματος στην ελλάδα. ήταν στην προεδρία σας που η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα κατά παράνομο τρόπο έκλεισε τις ελληνικές τράπεζες και δημιούργησε την απειλή χρεοκοπίας στην ελλάδα. ήταν κατά τη δική σας προεδρία που πετάξατε στα σκουπίδια τη βούληση του ελληνικού λαού που μέσα από ένα δημοψήφισμα με 62 αρνήθηκε την επιβολή νέου οικονομικού προγράμματο καταστροφή νέου μνημονίου είναι στη δική σα προεδρία που συνεχίστηκε η επιβολή ενό τέτοιου προγράμματο, δυστυχώ με την ανοχή σήμερα τη κυβέρνηση, που καταστρέφει την παραγωγική βάση τη χώρα, που πουλά τη δημόσια περιουσία και που εξαφανίζει κάθε ίχνος κοινωνικού κράτου στην ελλάδα. είναι στη δική σα προεδρία ότι χάθηκε κάθε ίχνος ανθρωπισμού καθώ συνεχίζονται να πνίγονται πρόσφυγε μετανάστες στο αιγαίο και στη μεσόγειο και εσείς δεν κάνετε απολύτως τίποτα. επομένως κύριε πρόεδρε του λουξεμβούργου και η δική σας προεδρία αποτελεί μια διάψευση όσων ελπίζουν ότι η ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στις αξίες της δημοκρατίας της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού και θέλω να σας πω ότι το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών δεν είναι μια τέτοια ευρωπαϊκή ένωση που έστω με αυτού του περιορισμένου ρόλου για έξι μήνε διευθύνεται δεν μπορεί να είναι το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών ούτε η φτώχεια ούτε η ύφεση ούτε ο ρατσισμό ούτε η μη διαχείριση των ανθρωπιστικών κρίσεων. σα ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. E ευχαριστώ Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε τα αποτελέσματα τη Λουξεμβουργική Προεδρία που θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω καταστροφική. Αυτοί οι έξι μήνε έφτασαν πρόσφυγε τρομοκράτε, αυξήθηκε ο φόβο και είχαμε τι επιθέσει στο Παρίσι και την Κολονία. Επ' αυτή τη Προεδρία παρέμεινε αδρανή η Ευρώπη. Στη δική μου τη χώρα, όποιο δεν κάνει τίποτα είναι συνένοχο. Ε, ε, ε, ξεκίνησε το σκάνδαλο των φορολογικών ελαφρύνσεων τη Λουξεμβουργική κυβέρνηση προ πολυεθνικέ. Όλοι ξέρουμε ότι η Επιτροπή Juncker έχει εμπλεχθεί σε αυτήν την ε, ε, ε, υπόθεση, εφόσον όταν ήταν πρωθυπουργό ο κ. Γιούνκερ ξέσπασε αυτό το είχε δημιουργηθεί αυτό το σκάνδαλο. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχνάμε αυτό το όνειρο σε αυτού του έξι μήνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αισθάνετε, κύριε Γιούνκερ, ντροπή και εσεί και όλοι οι συνάδελφοί σα για όσα έχουν γίνει. Έχουμε μπουχτίσει με την Ευρώπη των ισχυρών που παίζει το παιχνίδι των μεγάλων τραπεζών και των πολυεθνικών. Έχουμε αειδιάσει με αυτόν τον τρόπο σα. Και θα θέλαμε επιτέλου η Ένωση να ε, επιβραβεύει του ε, φιλό... τους έντιμου και φιλότιμου πολίτε χωρί να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη του. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών, ο κύριο Μαμίκιν τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές, είμαι από μια μικρή χώρα που πολλές φορές ε, από τους γείτονές που είναι πολύ ισχυροί, ξέρουμε και εμείς τι σημαίνει. Όπως και για το Λουξεμβούργο που είναι επίσης μια μικρή χώρα. Πάντως η Λουξεμβριανή Προεδρία έκανε πολλά για να βοηθήσει. Το προηγούμενο εξάμεινο λοιπόν ήταν σίγουρα ένα δύσκολο εξαιτία της επιδείνωση της μεταναστευτική κρίση και των επιθέσεων στο Παρίσι. Ελπίζω τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί να προστατεύσουν τα εξωτερικά μας σύνορα και να αποφέρουν καρπούς μακροπρόθεσμα. Τώρα, όσον αφορά το PNR και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Αυτά είναι από τα πιο θετικά αποτελέσματα που είχαμε το τελευταίο εξάμεινο. Θλίβομαι όμως που η δικιά μου χώρα, η Λετωνία, δεν μπόρεσε τα αποτελέσματα αυτά να τα προωθήσει πριν από το Λουξεμβούργο και χρειάστηκε να το κάνει αυτό το Λουξεμβούργο. Ευχαριστούμε. Η κυρία... Ο κύριος Άνεμανς. Ευχαριστώ. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώνονται όλες οι προεδρίες. Με συγχαρητήρια, με καλά λόγια, χτυπάμε στον νόμο, ε, λέμε ότι πόσο καλά πράγματα γίνανε. Όμως, μιλάμε μόνο για τις επιτυχίες. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει και άλλες επιτυχίες και άλλες επιτυχίες και άλλες επιτυχίες. Δεν μιλάμε για τις ε, αποτυχίες Λέμε ότι μπήκανε στο γρανάζι το θέμα της Φορολογικής Ένωσης, ενώ τίποτα για το LuxLeaks, τίποτα για άλλα ζητήματα. Μόνο συγχαρητήρια δίνουμε. Εδώ οι ευρωκράτες μπροστά σας συγχαίρουν και οι ευρωφανατικοί. Και το μόνο που λένε είναι ότι θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα περισσότερο το Συμβούλιο. Εγώ δεν θα πω τα ίδια κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Γιούγκερ, συνάδελφοι, ήθελα να ευχαριστήσω, σε αντίθεση με κάποιου άλλου συναδέλφου, τη Λεξουμβουριανή Προεδρία για την συνεργασία που είχε με το Κοινοβουλίο μα. Αλλά πάνω απ' όλα για την αφοσίωση και την προσοχή που έδειξε για θέματα καθοριστικά για το μέλλον τη Ένωση. Πάνω απ' όλα, ήθελα να σταθώ στη σημαντική στήριξη σε θέματα θεσμικού χαρακτήρα. Είδαμε πόσο στην Ευρώπη είναι σημαντικό όλο και περισσότερο να έχουμε ηγέτες που έχουν και τόλμη και μακροπνοία σχέδια και μια, ένα κοινό όραμα για το μέλλον μας. Αυτό το αποδείξατε για άλλη μια φορά από το Λουξεμβούργο και σας ευχαριστούμε. Ταυτόχρονα έγινε μεγάλο έργο για να εμβαθύνουμε την κοινωνική ένωση της Ευρώπης και να συμπεριλάβουμε κοινωνικές παραμέτρους στην οικοδόμηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ο στόχος αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμη πλήρω, όμως έχουν γίνει σοβαρά βήματα προόδου στη σωστή κατεύθυνση και υπολογίζουμε στην προθυμία σας για να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Τέλος, και νομίζω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά για να αποκτήσουμε όλοι κοινέ ευθύνε στο θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Ήταν ουσιαστική σημασία στα μέτρα και η συμφωνία του Ιουλίου ήταν ένα σημαντικό βήμα για να έχουμε μια κοινή πολιτική και σε αυτόν τον τομέα που η επόμενη Προεδρία θα πρέπει βεβαίως να περάσει στην υλοποίηση. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και νομίζω ότι θέλουμε μια Ευρώπη που να είναι χρήσιμη και όχι που να την επικρίνουν οι συνάδελφοι όπως κάνουν τώρα. Κύριο Σαρνέτσκι, ECR. Όχι. Και περνάμε στη διαδικασία Καρστιάη. Κύριο Φαπ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αξιολογήσω θετικά υπό τρεις ε, οπτικές γωνίες στη Λουξεμβουριανή Προεδρία. Καταρχάς, ε, σας αξίζουν συγχαρητήρια κύριε Πρωθυπουργέ και σε εσάς και στους υπαλλήλους σας για το μεγάλο θάρρος και την παρησία που επιδείξατε αναλαμβάνοντας ε, στην Προεδρία σας την ανάπτυξη δομών για τις διαγραμμικές δομές και τη διαγραμμική ασφάλεια βεβαίως με μια πολύ σημαντική βελτίωση που είχαμε εμείς επιφέρει στην πρόταση της Επιτροπής Μάλιστα σε περίοδο που δεν ήταν πρόεδρο τη Επιτροπή ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και γίνει αυτή η διόρθωση και μπορέσατε να δώσετε αυτή την προστιθέμενη αξία με του ευρωπαϊκού κανόνε για τι υποδομέ στο διαγραμμικό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο και συγχαρητήρια. Δεύτερον, στη φορολογική πολιτική που συζητήθηκε. Η Λουξεμβουριανή Προεδρία προχώρησε προώθησε τα θέματα αυτά και νομίζω ότι πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε πώς ε, αφενός μεν θα διαφυλαχθούν οι εθνικές προνομίες ως προς τη διαμόρφωση μιας φορολογικής πολιτικής αλλά ταυτόχρονα θα συνδυαστούν και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Μπορεί να έχουν διατυπωθεί βεβαίως από διάφορους επικρίσεις κατά του Λουξεμβούργου αλλά πρέπει να είναι ε, επιφυλακτικοί και προσεκτικοί αυτοί οι οποίοι ε, ίσως μια μέρα δουν την ε, Ιρλανδία να κατηγορείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απουσία αλληλεγγύης ευρωπαϊκής και όχι φορολογικές παραβάσεις. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι για τη δυνατότητα που είχαμε να συναντηθούμε και στις Βρυξέλλες με τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Λόπες Αγουίλαρ. Στη συζήτηση αυτή αναφερθήκαμε στα επιτεύγματα της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Δεν μιλήσαμε όμως αρκετά για τα θέματα εκείνα τα οποία μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε, που βρίσκονται στο Συμβούλιο εδώ και χρόνια. Η οδηγία, για παράδειγμα, για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ποινικού δικαίου. Δυστυχώς το Λουξεμβούργο δεν κατάφερε να ξεμπλοκάρει το θέμα αυτό. Το στοιχείο κλειδί είναι η συζήτηση όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας ενώ η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι πρόκειται για κύριο πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο δεν συμφωνεί. Και χρειάστηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που βγήκε το Δεκέμβριο και λέει ότι απάτε σε βάρο των δημοσιοκών συμφορέντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο των χωρών μελών. Αυτό πρέπει να επηρεάσει την οδηγία ΠΙΦ για τα δημοσιονομικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν μέσα σε αυτή τη δυναμική του τρίο που έχει η Ολλανδική Προεδρία τώρα με τις επόμενες, η οδηγία αυτή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεμπλοκαριστεί και να προχωρήσει. Ευχαριστούμε κύριο Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, ο χειρισμός του προσφυγικού από την Λουξεμβουργιανή Προεδρία είναι μνημείο αποτυχίας, αφού με τους χειρισμούς της μετέτρεψε την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες βρίσκονται πλέον στα νησιά του αιγαίου και στις υπόλοιπες περιοχές της ελλάδας. η πολιτική της περίφημης πεντεγκατάστασης των 160.000 προσφύγων έχει αποτύχει κύριε πρωθυπουργέ του λουξεμβούργου έχει αποτύχει κύριε γιούνκερ. μόνο οι πρόσφυγες έχουν μετακινηθεί με το σύστημα αυτό μέχρι το δεκέμβριο υπολογιζόταν σε 184. τι γίνεται με την τουρκία; θοπεύετε την τουρκία γιατί είναι γνωστό ότι η τουρκία και η τουρκική ηγεσία ενθαρρύνει τα δουλεμπορικά κυκλώματα και δεν έχετε πάρει μέτρα απέναντι σε αυτό και υπάρχουν καταγγελίες και έχουμε στοιχεία. ταυτόχρονα με την προώθηση της νέας frontex αυτό που κάνετε είναι να δημιουργείτε ένα μηχανισμό όπου θα έχει δυνατότητα επιχειρησιακής επέμβασης και δράσης πάνω από τη θέληση και των κρατών και των κυβερνήσεων και αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδος και τη μετατρέπει αυτόματα σε προτεκτοράτο. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Μπετέλ, κύριε Γιούνκερ. Προέρχεστε και οι δύο από χώρα διαπνεόμενοι από το κοινοτικό πνεύμα και αγωνιστήκατε ώστε να προχωρήσει και στην καταπολέμηση τρομοκρατίας όπου ήταν πολύ σημαντικό το θέμα του PNR, του καταλόγου ε, ονομάτων επιβάτων πτήσεως ε, αλλά θέλω να ρωτήσω, δεν νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο και επιτέλους να υπάρξει μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των ευρωπαϊκών κρατών και ένα θέμα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είχαν κρίνει ως απολύτω ε, πρώτης προτεραιότητας οι Αμερικανοί μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Τώρα φαίνεται να το επισημαίνει μόνο η Γαλλία ως ζήτημα προτεραιότητας. Το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τσάτρα-πάτρα. Βεβαίω και είναι ένα καταπληκτικό όπλο στα χέρια των τρομοκρατών το θέμα της χρηματοδότησης, τα κονδύλια που μπορούν να ε, διακινούνται. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ αυτόν, ε, αυτή τη σκητάλη θα την παραδώσετε στην Ολλανδική Προεδρία κύριε Μπέτλ και εσείς κύριε Γιουνκέρ είστε διατεθειμένος να προωθήσετε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Σας ευχαριστώ. Δεν περιμένω να μου δώσετε το λόγο. Θα τα πω στα αγγλικά. Πολλές φορές τα ακριβά αρώματα έρχονται και σε μικρά μπουκάλια. Αυτό ισχύει για τους ανθρώπους αλλά και για τις χώρες. Και ε, το Λουξεμβούργο ήταν για πολλωστή φορά σε κεντρικό ρόλο και καθοδήγησε πολύ σωστά τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ε, συγχαίρω λοιπόν για το εξαιρετικό σας έργο τους τελευταίους έξι μήνες ε, και για την πρόοδο που επιτελέσατε και τρεχαστήκατε πολύ αποτελεσματικά, ήδη στον τομέα που με ενδιαφέρε εμένα, δηλαδή την ε, προστασία των πολιτών και συμμετείχα σε πολλούς τριμερείς διαλόγους. Και πρέπει να πω ότι ο πρόσωπο σας από το Συμβούλιο ήταν πολύ δίκαιο δίκαιος, σταθερός, αξιόπιστος και ε, δραστήριος. Ε, ε, πετύχαμε να ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματος αυτού. Υπήρχε μια πολύ καλή έκβαση και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα κανονισμός που πετύχαμε. και η πρώην Επίτροπος Ρέντινγκ που είναι από το Λουξεμβούργο και που ήταν η εμπνεύστρια αυτής της πρότασης είναι, και επίσης και εκείνη την ευχαριστούμε για τη δουλειά της. Ο κύριος Φουντούλη. Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας, θέλω να πω ότι οι μη εγγεγραμμένοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν εκλεγεί με διαφορετικό τρόπο από όλους τους άλλους συναδέλφους. Δυστυχώς, κατά τη διαδικασία του Catch the Eye, ποτέ δεν παίρνουμε χρόνο ομιλίας. Ήδη ο χρόνος μας, σαν μη εγγεγραμμένοι, είναι πολύ περιορισμένο Και έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι να παίρνουν από τις πολιτικές ομάδες το λόγο στο ΚΑΤΣΔΙΑΙ και εμείς να είμαστε αποκλεισμένοι. Σας ευχαριστώ και πρέπει να επιληφθείτε του θέματος. Δεν είχαν ζητήσει τη στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΙ μία εγγεγραμμένη βουλευτές. Εξ αυτών ο κύριος Μπάλτσο έλαβε το λόγο νωρίτερα. Από αυτούς που είχαν ζητήσει δηλαδή. Ο κύριος Μαυρίδης έχει το λόγο. Thank you, Mr. President. Uh, Ευχαριστώ. Θα έχουμε παρατηρήσει τους τελευταίους μήνες. Τι έχουμε δει λοιπόν τους τελευταίους μήνες. Την επιμονή του Ερτογάν στην Τουρκία να μην εφαρμόζει τις υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, συνεχίζει την κατοχή της Κύπρου και συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά των ίδιων των Τούρκων. Ακαδημαϊκοί διώκονται, Κούρδοι στις κουρδικές επαρχίες της Τουρκίας κλπ. κλπ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή. Πιστεύετε, και αυτό έχει να κάνει με την ίδια την Επιτροπή, Πιστεύετε ότι οι πολιτικές μας απέναντι στον Ερτογκάν τους τελευταίους μήνες ήταν αποτελεσματικές. Βασίζονται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ηθική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βασίζονται σε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία Καριστιά, κυρίε και κύριοι, και περνούμε στον κύριο Γιουνκέρ εκ μέρου Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα πάρα πολλές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα περιοριστώ λοιπόν σε αυτές που με αφορούν γιατί οι περισσότερες παρατηρήσεις ήταν θετικές, αφορούσαν την κυβέρνησή μου και έχω βέβαια το την ευτυχία να ε, μην χρειάζεται σήμερα, κάτι εξαίρεση, ε, να κάνω πολύ λεπτομερείς ε, απαντήσεις. Θα απαντήσω λοιπόν στις δύο-τρεις ερωτήσεις που απευθύνθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως εκείνη που έχει να κάνει με τη συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Δεν προχωράμε πραγματικά. Από ό,τι φαίνεται, οι μυστικές υπηρεσίες είναι τόσο μυστικές που δεν βλέπουμε καν με ποιον τρόπο συνεργάζονται. Ήδη το 2001, όταν είχαμε τα γεγονότα της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, τότε υπό τον Κίφερ Χόστατ το Συμβούλιο είχε πάρει κάποια μέτρα για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των χωρών μελών της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά δεν έγινε περίπου τίποτα. Στη συνέχεια, μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν και που έφτασαν ως εμάς, ότι υπήρχαν λήψεις σε θέματα συνεργασίας μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών και μεταξύ των αστυνομικών αρχών, είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε μία παραπάνω προσπάθεια. Δεύτερον, Μας ρωτήσατε για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσης το Φεβρουάριο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρωθυπουργός Μπέτλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο για το θέμα της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Πρώτο θέμα τα ερωτήματα που τέθηκαν για τις σχέσεις με τον Ομένο Βασίλειο. Βρισκόμαστε σε θέση αναμονής για ένα τελικό κείμενο. Δεν είναι αρμοδιότητα της εξαμηνίας προεδρίας. Ο πρόεδρος Τούσκ θα πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την ε, Βρετανική κυβέρνηση. Οπότε δεν θα επεκτάθω. Κύριε Παπαδημούλη, μιλήσατε για κάποια προβλήματα, ε, όπως και άλλοι συνάδελφοι, προβλήματα μετανάστευσης και συμφωνώ, δεν, είναι μονόδρομοι, δεν πρέπει να είναι μονόδρομοι η αλληλεγγύοι. Πρέπει οι δεσμεύσεις και των ε, μεν και των δε να γίνονται σεβαστές. Το κόστος σήμερα έχουμε την εντύπωση ότι τεπομίζεται κυρίως η Ελλάδα. Όμως και η Γερμανία, κάθε χώρα προορισμός ε, έχει κόστος να αναλάβει. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε μία χώρα. Πρέπει όμως επίσης να πούμε σήμερα ότι τα hot spot δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τους Έλληνες ε, συναδελφούς μας για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Δεν αφήνουμε μόνο της την Ελλάδα. Η Ελλάδα και οι άλλες χώρες που ε, έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι το Λουξεμβούργο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ω προ το Σύμφωνο Σταθερότητα ζήτησε ε, αλλαγή στι δαπάνε, ευελιξία στι δαπάνε για να καλύψουμε και το θέμα τη ε, Η κυρία Λεπέν ήρθε στις 9.40 και έφυγε στι 9.45, οπότε δεν μπορώ να τη απαντήσω, εφόσον δεν βρίσκεται εδώ και ως προς τις παρολογικές συμφωνίες. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία θα μπορούσε να πάει παραπέρα πιο μακριά για όλες τις φορολογικές συμφωνίες και αυτές που είναι αποκλειστικά εθνικού χαρακτήρα. Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για το Λουξεμβούργο είναι όροι που δεν αξίζουν καν να το σχολιάσω. Η κυρία Μπερές, μιλήσατε για τη χρηματοδότηση της θερμοκρατίας. έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είναι προτεραιότητα για το 2016 και το Λουξεμβούργο θα στηρίξει αυτή την προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά το Μητρό Επιβατών, πράγματι το είπε και ο πρόεδρο Γιούγκερ μόλις τώρα, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών και θα πρέπει να ενισχυθεί. Το συζητάμε, είναι καιρός να προχωρήσουμε. Και σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Λόπε Αγγιλάρ, ναι, θα πρέπει η απάτη, η φορολογική απάτη, να είναι ποινικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ευχαριστήσω για του επένου σας προ την κυβέρνηση και του συνεργατέ τη. Σίγουρα κάποιοι θα θέλουν να έχουμε προχωρήσει παραπέρα, πιο μακριά, κάποιοι θεωρούν ότι ήδη ξεπεράσαμε τα όρια. Όμω, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε σήμερα και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα κύριε Πρόεδρε, να το αναγνωρίσουμε και είναι είναι γέφυρες μεταξύ των ε, ε, πολιτισμών, των θρησκειών, των ανθρώπων, των χωρών και αυτές θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε για το καλό της Ένωσης και για το μέλλον. Ελπίζουμε και κάτω να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστούμε.